Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ, οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Αυστρία. Α, ο κύριος Χάουιτ έχει ένα διαδικαστικό. Κύριε Χάουιτ, έχετε το λόγο. διαδικαστικό με βάση το άρθρο 96. Θα ήθελα να, ρωτήσω, να ζητήσω από την Πρόεδρο να στείλει επιστολή στην, στην ομάδα της Φόρμουλα 1 γιατί για λογιστικούς λόγους δημιούργησαν ε, πρόβλημα στη διοργάνωση της ε, Φόρμουλα 1. Θα ήθελα να υπεθυμίσω ότι υπάρχει ε, α, υπάρχουν τέτοια προβλήματα που εμποδίστηκαν ε, από συμμετοχή, σημαντική αποσυμμετοχή σε αθλητικούς ε, αγώνες ή σημαντικές αθλητικές ε, οργανώσεις. Αν κάποια ομάδα αποσύρεται για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να τύχουν της υποστήριξής μας και το αιμοβόρο όνομα του Μπαχρέιν δεν θα πρέπει να στέκεται φέτος δίπλα στα υπερήφανα ονόματα των ευρωπαϊκών ομάδων. Όνουμε το θέμα αυτό κύριε Χόουιτ. Σας ευχαριστώ για την επεσήμανση. Θα την ε, μεταφέρουμε. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν την... Α, και άλλο διαβιβαστικό, και άλλο ναι, διαδικαστικό. Ο κύριος Λίτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο εισηγητής της έκθεσης για τις συμφωνίες διμερών ε, επενδύσεων για τη μεταβατική περίοδο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά προσεκτική ανάλυση της, ψηφο... ανάλυση ψηφοφορίας ε, στο Κοινοβούλιο και της πρότασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα ήθελα να αποσύρω το όνομά μου από την έκθεση αυτή γιατί το Συμβούλιο... η θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι μονομερός υπέρ των επενδυτικών συμφερόντων και δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη την ανάγκη για διαφάνεια. Και τα παλιά κράτη-μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των νέων χωρών μελών υπάρχει μια ισορροπία. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των επενδυτικών συμφερόντων και των περιβαλλοντικών και νομικών κριτηρίων. Δεν μπορώ λοιπόν να υπεραμηθώ τι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θέλω να είμαι επικεφαλή των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να αποσύρω το όνομά μου και να αφήσω την έκθεση αυτή στην Προεδρία τη Επιτροπή. Καστικό και πρέπει να το αφαίρετε στην αρμόδια Επιτροπή. Ε, Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να είστε ακριβεί στον χρόνο, διότι καταλαβαίνετε είναι μέρα ε, ψηφοφοριών και αναχώρηση των βουλευτών στη συνέχεια και δεν πρέπει να καθυστερήσουμε να πάμε στις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Ερχόμαστε στο θέμα σήμερα της ε, ημερήσιας διάταξης. Θα ξεκινήσουμε με τον ε, εισηγητή τον κύριο Βίλαντ. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Μιλώ εξ ονόματο τη κυρία Ματζόνη, Προέδρου τη Επιτροπή μα, η οποία δυστυχώ δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα στην Ρωμέλεια και σίγουρα υπάρχουν πιο σημαντικέ αναφορέ από την προκείμενη. Στην αναφορά αυτή δεν έχουμε 30.000 θύματα όπω σε άλλε αναφορέ. Πρόκειται για τη φύση, για την τοπική οικονομία, για την δυνατότητα ανάπτυξη. Αυτά διακυβεύονται. Και Μιλάμε για την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία μικρή παρατήρηση εκ των προτέρων. Επιτρέψτε μου η αναφορά για το θέμα αυτό, για την υπόθεση αυτή, για τους αναβατήρες αυτούς, καταδεικνύει ότι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αρέσκονται να ρίχνουν λάσπη στο μεν ή στους δε. Ο ένας είναι για την φύση, ο άλλο για την οικονομία, οι τοπικέ αρχές, η τοπική κυβέρνηση. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ενδείκνυται η υπόθεση για τέτοια λασπολογία. Ε, η κυρία Λέχτενμπέργκερ ε, παραβρέθηκε σε μια αποστολή διερευνητική εκεί μαζί μου και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να αποτελεί μια εποπτική αρχή. Αυτό είναι καταδεικνύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πρέπει να αφήσουμε όμως ε, την, τις εργασίες και τις αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές. Οι αναφέροντες ε, ανέφεραν ότι δεν τηρήθηκε το όριο των 20 εκταρίων και ότι καταθμήθηκε τεχνητά το έργο σε ε, μικρότερες εκτάσεις για να μην χρειαστεί η διεξαγωγή μελέτης αντικτύπου, μελέτης επιπτώσεων. Εν τω μεταξύ έχει μετατραπεί αυτό το όριο σε 10 εκτάρια, άρα έχει τροποποιηθεί η κατάσταση. Μεταβήκαμε λοιπόν επιτόπου και διαπιστώσαμε ότι οι διατάξεις ε, οι οποίες ε, προκύπτουν από τον κανονισμό για το περιβάλλον είχαν τηρηθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου στην Αυστρία. Μπορούμε φυσικά να ε, ζητήσουμε διευκρινήσεις για ένα τετραγωνικό μέτρο, για ένα μέσο ή οτιδήποτε, αλλά δεν θεωρούμε ότι καταφανώς ε, θα έπρεπε να καταδικαστεί το έργο σε ό,τι αφορά λοιπόν τα τμήματα και ούτω καθεξής του έργου. Αλλά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε ενδελεχέστερα τη συγκεκριμένη κατάσταση και το θέμα ήταν αν κατά πόσο Ήταν σωστή η στάση της πρωτεύουσα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παρατηρούμε λοιπόν τέτοια φαινόμενα όχι μόνο στην Αυστρία, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη και στο δικό μου κράτος μέλος. Πώς γίνονται αντιληπτές οι δυνατότητες διαμόρφωσης. Ανακύπτει το ερώτημα το κατά πόσο θα πρέπει να επιτρέπεται η τοπική κατάθμιση των έργων ή η χρονική κατάθμιση των έργων για να διευκρινιστεί δηλαδή κατά πόσο ε, ένα έργο αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου έργου, ετεροχρονισμένο. και από πλευράς νομικής διαμόρφωσης εάν υπάρχει κατάθμιση έργων. Και το θέμα είναι πώς οι ευρωπαϊκές διατάξεις ε, επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν η θελημένα ή μη την κατάτμιση αυτή και κατά πόσον θα πρέπει να καταστούν πιο αυστηρές. Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε οι πίστες σκι ενός, δύο, δέκα εκταρίων οι οποίες ε, διευρύνονται να μένουν εκτός των υπολογισμών. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκές διατάξεις προβλέπουν ότι τα μεγάλα αυτά έργα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη συνολική ωφέλιμη έκταση. Και θέλουμε να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αντιμετωπίζει το θέμα. Κύριε Βίλαν, ήσασταν και πολύ ακριβή στον χρόνο. Τώρα ο κύριος Σότιγκερ θα πάρει το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mr. Commissioner, you have the floor. Αξιότιμες ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαιρόμαστε ως νόβληφος Πότνα και εγώ που έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο έχει την εποπτεία όλων των περιβαλλοντικών διατάξεων και η οδηγία αυτή έχει μεγάλη αξία στη συγκεκριμένη περίπτωση στην οικονομική και οικολογική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί για μας ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Τα έργα τα οποία είναι σημαντικά σε, ως προς την επίπτωσή του στο περιβάλλον πρέπει να υποβάλλονται σε μια μελέτη αντικτύπου, σε μια μελέτη επιπτώσεων, προκειμένου να διευκρινιστούν οι έμεσες και άμεσες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Μιλάμε για έργα και ίδια εργών, όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει βάσει οριακών τιμών να αποφασίσουν κατά πόσον χρειάζεται τέτοια μελέτη επιπτώσεων. Η περίπτωση της δικής σας περιοχής συγκαταλέγεται σε ένα είδος έργων όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει αν επιτρέπονται καν τα έργα. Αν επιτρέπεται καν η διεξαγωγή έργων. Η αυστριακή νομοθεσία δεν ήταν αρκετά ικανοποιητική στο παρελθόν. Μιλούσαμε για 10 εκτάρια ή για 20 εκτάρια και άνω. Ε, αφού του την ε, αναφορά, απευθύναμε έτοιμα προς την Αυστριακή Κυβέρνηση ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς ε, ε, εφάρμοσε τη σχετική οδηγία. Μας απάντησε η Αυστρία ότι δεν είχε γίνει μελέτη επιπτώσεων δεν ήταν απαραίτητη γιατί δεν είχε ε, ξεπεραστεί η οριακή τιμή των 20 εκταρίων. Υπήρχαν και εκφράστηκαν επίσημες αμφιβολίες εξ ονόματός μας και διαπιστώσαμε ότι για τον ορισμό της ε, έκτασης του έργου και προκειμένου να, προκειμένου να αποφασιστεί αν χρειαζόταν μελέτη επιπτώσεων δεν ε, πρέπει να λεφτεί μόνο η υπόψη η περιοχή με την στενή της έννοια και στη συνέχεια η Αυστρία και αυτό πιστεύω είναι η σημαντική συνέπεια της αναφοράς αυτή, αυτής, ε, ανανέωσε, ενημέρωσε την σχετική νομοθεσία για να συνάδει με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η απόφαση για το κατά πόσο είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μελέτης επιπτώσεων εξαρτάται πλέον από το εύρος της διεύρυνσης της περιοχής ε, της πίστας σκι και από την ε, έκταση, την, την, την στην οποία διεξάγεται. Είναι λοιπόν πλέον σαφής η νομοθεσία και αυστηρής η νομοθεσία για τη μελέτη εκτάσεων, επιπτώσεων. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα κατακαιρματισμού των έργων ελέγχουμε και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, το θέμα των επιπτώσεων στην ε, φύση. Και διευκρινίστηκε ότι σκοπός της οδηγίας ΕΠΕ δεν είναι να υπάρχει δυνατότητα ε, να καταργηθεί αυτή η ανάγκη εξέτασης του συνόλου του έργου. Το θέμα είναι τα κατασκευαστικά μέτρα και το πώς εντάσσονται στην όλη περιφέρεια. Άρα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα μέσα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του έργου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη ε, έκταση πριν από τη διεύρυνση θα έπρεπε να έχει γίνει screening, έλεγχος για να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν απαραίτητη η διεξαγωγή μελέτης επιπτώσεων για το έργο. Και αυτό το αποτέλεσμα θα έπρεπε να έχει δημοσιευθεί. Οι αυστριακές αρχές δεν ε, εκπληρώσαν αυτές τις υποχρεώσεις τους, δεν κάναν το σχετικό screening, το οποίο θεωρούμε ότι προδιαγραφόταν από την νομοθεσία. Το έργο πλέον ε, ανήκει στο παρελθόν εγκρίθηκε και, και αποφασίστηκε πριν από πέντε χρόνια, έχει ολοκληρωθεί η οικοδόμησή του, η κατασκευή του. Λάβαμε ε, λεπτομέρειες, ε, ζητήσαμε μάλλον λεπτομέρειες από τις σχετικές αρχές για τις ε, ενδεχόμενη ανάγκη αποδυνάμωσης, αν θέλετε, των επιπτώσεων. Θα ελέγξουμε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες και βάσει των πληροφοριών αυτών θα δούμε κατά πόσον μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω μέτρα για την ε, μείωση των επιπτώσεων στη φύση. Ζητήσαμε από τις Αυστριακές Αρχές να μας επιβεβαιώσουν ότι σε τεχνητές διευρύνσεις και της συγκεκριμένη ε, περιοχής αλλά και άλλων περιοχών σκι θα συμβαίνει πάντα καταρχάς ένα screening προκειμένου βάσει του ελέγχου αυτού να αποφασίσετε αν χρειάζεται διεξαγωγή ή μη μελέτης επιπτώσεων. Ο συνάδελφος Ποτότσνικ βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας ε, αναθεώρησης της οδηγίας ΕΠΕ. Θα υποβάλει ένα νέο κείμενο το οποίο θα δίνει πιο μεγάλη ε, έμφαση σε θέματα φυσικής, ε, φυσικών επιπτώσεων, θα δίνει βάρος σε θέματα βιολογικής θα συμπεριλαμβάνει την απόφαση του ΔΕΚ και θα αποκλείονται ακόμα πιο αυστηρά δυνατότητε παράκαμψης της οδηγίας. Βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας λοιπόν της ε, νέας αυτής ε, μορφής της οδηγίας και έχει διεξάγει διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 2012 θα, υποβάλλεται θα υποβάλει σχετική πρόταση, το αργότερο, και κατά κανόνα οι καταχρηστικές αυτές εφαρμογές ε, της οδηγίας θα βελτιωθούν προκειμένου, προκειμένου να μην υπάρχει δυνατότητα παράκαμψης ε, της νομοθεσίας. Χαιρόμαστε που η οδηγία ή μάλλον η νομοθεσία στην Αυστρία πλέον συνάδει με την οδηγία ΕΠΕ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι κατά τη μελλοντική διεύρυνση των ε, περιοχών αυτών για σκι ε, θα εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άρα όλοι έχουμε μάθει από τα παθήματα αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης κύριε επίτροπε ευχαριστώ πολύ. τώρα ερχόμαστε στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. ξεκινάμε με την ομάδα του ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος ο κύριος Ζάρ για δύο λεπτά. κρατήστε τον χρόνο σας παρακαλώ κύριε συνάδελφοι είμαστε ήδη με καθυστέρηση. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, ο συνάδελφος Βίλαν θα παρουσίασε το περιεχόμενο με σαφήνεια, το περιεχόμενο της υπόθεσης. Θα ήθελα να κάνω κάποιες πολιτικές εκτιμήσεις. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, το γεγονός ότι ελέγχουμε την ε, εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ. Γιατί πάντα υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών οδηγιών και της μεταφοράς σε εθνικό επίπεδο. Δεν είμαστε αναθεωρητικό όργανο στην Επιτροπή μας, αλλά θεωρώ ότι είναι γεγονός ότι βλέπουμε από τη συγκεκριμένη αναφορά ότι γίνεται διαφορετική ερμηνεία των ευρωπαϊκών οδηγιών σε εθνικό επίπεδο και τελικά η αναφορά αυτής οδήγησε στην τροποποίηση μια νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία και είμαι περήφανο γι' αυτό. Θεωρώ την επιτυχία τη ευρωπαϊκή πολιτική. Κατά δεύτερον, το πρόβλημα το οποίο διακρίνω γενικά και αυτό το απευθύνω και ως ερώτηση προς τον Επίτροπο. Διαρκώς βλέπουμε ότι πάρα πολλοί πολίτες ασχολούνται με την εφαρμογή ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου στην, ε, σε εθνικό επίπεδο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ε, πρόκειται για νομοθεσία και σε εθνικό επίπεδο. Και όταν ε, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφανθεί για κάποιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ε, της υπόθεσης, μας λένε ότι το χύψη κρατος μέλος εφαρμόζει κατά το δέον τρόπο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν υπάρχει λόγος παρέμβασης. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα μέσο προκειμένου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όταν διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διάλογο με το κράτος μέλος που ε, εμπλέκεται. Γιατί πλέον στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε λύσει για το μέλλον, αλλά όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών, ο κύριος Για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη εδώ μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα μάθημα για το μέλλον. Εμείς οι Αυστριακοί είμαστε ε, υπέρμαρχοι του σκι. Πώς να το κάνουμε. Και χρειαζόμαστε και πίστες σκι. Αλλά στις πίστες ε, στο σκι χρειάζεται, για να κάνουμε σκι χρειάζεται και ένα όμορφο περιβάλλον. Ιδάλλως τι νόημα έχει το σκι. Και ότι από τη συγκεκριμένη κατάσταση η αυστριακή πολιτική, μάλλον νομίζω θεωρώ ότι και στο μέλλον έχει κάνει πολλά σφάλματα. Μονομερή ε, έργα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον είναι βιώσιμα αυτά τα έργα και αυτό ήταν και η πρακτική της διοίκησης. Έτσι ήταν τα πράγματα και εδώ διακρίνουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πράγματα πήγαν στραβά από ό,τι φαίνεται και σε πολλέ περιπτώσει, όταν πηγαίνουν στραβά τα πράγματα, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση κατατέθηκε μία αναφορά. Υπήρξε μία αντίδραση. Και τα πράγματα ε, βελτιώθηκαν στην Αυστρία και νομίζω ότι αποτελεί ένα καλό υπόδειγμα του πώ πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Για την ομάδα των Πρασίνων, η κυρία Λίχτεμπεργκερ για ένα λεπτό επίση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες σας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Εγώ θα ήθελα μόνο μία επερώτηση να κάνω. Είπατε ότι σε ό,τι αφορά ε, την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ, ε, πλέον η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη σε ό,τι αφορά την Αυστρία. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία ε, ελέγχου, κατά πόσο χρειάζεται διεξαγωγή μελέτης αντικτύπου, θα θέλαμε να υπάρχει συμμετοχή και των πολιτών προκειμένου να υπάρχει ένα σύστημα έγκριση προειδοποίησης και να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο όπως ε, στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Το πολύ σημαντικό για μένα είναι να μην συμπεριλαμβάνονται και να μην, ε, μάλλον το να μην ε, συνυπολογίζονται οι πίστες διεύρυνσης, μάλλον να συνυπολογίζονται σαν ξεχωριστέ περιοχές και εκτάσεις όταν έχουμε σκάψει όλο το βουνό, ε, θεωρώ ότι αυτό είναι παράλογο. Ελπίζω ότι συγκεκριμένη περίπτωση θα την λάβουμε υπόψη και στο μέλλον για τις μελλοντικέ διαδικασίες. Για δύο λεπτά από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ έχουμε μία περίπτωση που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ρυθμίσουμε κάτι που όντως αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έθεσε ο κύριος Γιάρ και θα συμπεριλάβουμε στην ετήσια μας έκθεση που θα, θα υποβάλει η Επιτροπή Αναφορών για το 2010. Μπορεί ε, το Μελάο Ντάνιμς να μας χρησιμεύσει ως παράδειγμα και στα Πυρηναία και στις Άλπεις, γιατί το γεγονός ότι υποβάλλεται αναφορά από Ευρωπαίους πολίτες, από τη στιγμή που υποβάλλεται μέχρι να διεκπαιρεωθεί το θέμα, περνάει τόσο καιρός μπορεί να δημιουργηθεί ένα επανόρθωτη ζημία. Θα πρέπει αυτό να μας γίνει μάθημα. Γιατί υπάρχει κοινοτική οδηγία που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να πραγματοποιήσουν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα σε ευαίσθητες από οικολογική απόψη περιοχές όπως είναι οι Άλπεις, όπως είναι ε, τα Πυρηναία στην Ισπανία. Για να παραγωνιστεί η οδηγία, στην περίπτωση αυτή κατατμήθηκαν οι περιοχές για να αποφευθεί υποχρέωση ε, κατάρτισης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά η ΕΠΕ. Αν όντως το πιστεύετε αυτό, θα πρέπει να, δρά, να δράσετε ε, πολύ πιο άμεσα από τη στιγμή που υποβάλλονται αναφορές σε καταγγελίες ε, και για έργα που χρήζουν μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει να μην αφήνουμε τόσο χρόνο να περνάει. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντηρηθούν αυτές οι προθεσμίες και να μην μπορούν τα κράτη-μέλη να παραμερίζουν ε, την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ, γιατί πολλές χώρες το έκαναν, όχι μόνο η Αυστρία και η Ισπανία. Έχουμε ένα κρεμές έργο στα Πυρηνέ και πάλι για χιονοδρομική πίστα στην Παιδιάδα Καστανέσε και το ίδιο θα κάνει και η Ισπανία. Η αρμόδια αρχή θα κατατμήσει αυτό το έργο για να εμποδίσει ναι, να παρακάμψει αυτή την υποχρέωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμε κύριε Επιτροπέ ΕΡ. Σκοπός της οδηγίας ΕΠΕ είναι σύμφωνα με τις αρχές που επικρατούν να μελετηθούν οι άμεσες και έμεσες επιπτώσεις των έργων. Η παράκαμψη έργων που έχουν ωστόσο σχέση με τέτοια μεγάλα έργα οδηγεί ε, νομοτελειακά σε υπονόμευση της οδηγίας αυτής. Γι' αυτό αποφασίστηκε λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο σκοπός της οδηγίας δεν είναι η κατάτμιση και η παράκαμψη έτσι της οδηγίας από τα κράτη-μέλη. Και το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν ε, ήταν ε, η εθνική νομοθεσία αυτή που παρουσίασε προβλήματα, αλλά η πρακτική εφαρμογή και μία σύσταση τότε ήταν προς τα κράτη-μέλη και ορίστηκαν οριακές τιμές όπως και την Αυστρία. Συστάθηκε στις χώρες να διεξάγουν ένα κατάλληλο screening, ένα έλεγχο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ευαίσθητες περιοχές μέσω συσσόρευσης των έργων. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Οι Αυστριακοί πολίτες ε, σε πολλές περιπτώσεις έχουν διαμαρτυρηθεί και έχουν ε, δηλώσει ότι δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη τα δικαιώματά τους και τα συμφέροντά τους. Θα πρέπει η εθνική νομοθεσία να είναι αρκετά ενδελεχής για να προβλέπει τέτοιες περιπτώσεις. Πώς εκτιμάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη στάση της Αυστρίας και την Αυστριακή νομοθεσία. Η κριτική για την έλλειψη συμμετοχής των ε, πολιτών στη διαδικασία αυτή ισχύει για όλα τα κρατημέρια λίγο πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να ερευνηθεί και η ενιαία ε, διαδικασία για τη συμμετοχή των πολιτών στην συζήτηση. Ερχόμαστε τώρα στον κατάλογο των άλλων εγγεγραμμένων μιλητών. Ο κύριος Σίμπερ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι ο κατάλογος των ομιλητών καταδεικνύει ότι θεωρείται ως ε, ε, ανώτερη αρχή η Επιτροπή Αναφορών. Μιλάμε για ένα έργο για δύο μικρές κοινότητες στην Αυστρία. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε με τον καλύτερο τρόπο να εφαρμόσουμε την αυστριακή νομοθεσία και νομίζω ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τις αρχές της Αυστρίας για οποιαδήποτε σφάλμα. Το θέμα είναι να έχει εφαρμοστεί σωστά η οδηγία ΕΠΕ στην Αυστρία και να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές νομοθετικές παραδόσεις στην Αυστρία και στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Νομίζω ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας προσπάθησε να μεταφέρει σωστά την, ε, την νομοθεσία. Εκ των υστέρων οι νομομαθείς κατέληξαν στο ότι μπορεί να παρουσιάστηκαν σφάλματα, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι μιλάμε για ένα τελευταίο ποσοστό το οποίο συζητάτε. Έγινε και μεγάλες πληρωμές και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια πολιτική εκτίμηση εκ των υστέρων λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο αυτό προσπάθησε να κάνει μια εξυγίανση των όσων έχουν συμβεί. Νομίζω ότι έχει μια πράσινη σφραγίδα. Θα πρέπει να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο αυτό να κοιτάξει και εκτός των συνόρων. Να κοιτάξει και οι υποθέσεις όπου το ποσοστό σφάλματος του κράτους μέλους είναι πολύ πιο υψηλό. Θα πρέπει λοιπόν να τα λάβει όλα αυτά η υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στην περιβαλλοντική πολιτική. Πολύ κύριε Σύμπε. Ο επόμενος εγγεγραμμένος ομιλητής, ο κύριος Μόλζερ, δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα, οπότε ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο <clears throat> τέσσερις συνάδελφοι και ο κύριος Βίλαν θα πάρει το λόγο στο τέλος όμως για να ακούσει και τους άλλους συναδέλφους. Ε, ο κύριος Μπέκερ, για ένα λεπτό παρακαλώ, οι παρεμβάσει κάτω στη Ο κύριος Μπέκερ. Ε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμοι επίτροπε, θα ήθελα να αναφέρω και να τονίσω αυτό που είπε ο Επίτροπος, ότι έμαθαν οι εθνικές αρχές, γιατί νομίζω ότι η υπόθεση αυτή της αυστριακής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τον ε, Υπουργό Περιβάλλοντος ε, θα πρέπει να εξελογηθεί θετικά λόγω της τροποποίησης της εθνικής ε, νομοθεσίας και θα πρέπει να θεωρηθεί και να αναφέρεται ως υπόδειγμα για πολλές άλλες περιπτώσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν πολλοί κόσμος. Αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Γιάρ. Ο σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες ε, τιμές, συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα, θα χρησιμοποιούνται στην αρχή και στο τέλος ενός έργου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερέρα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα σύντομα σχόλια μετά από αυτή τη διαδικασία. Η εμπειρία της έμπρακτης εφαρμογής της διαδικασίας τη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρά τις θετικέ πτυχές που περιλαμβάνει μας δείχνει ότι ε, επιδέχεται βελτιώσεων. Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στις ε, αναλύσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γιατί πολλές φορές ε, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος και χανόμαστε τις λεπτομέρειες και χάνουμε τη γενικότερη προοπτική. Θα πρέπει να δούμε με πιο σφαιρικό τρόπο τον χαρακτήρα των ανθρώπινων επιπτώσεων στη φύση θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον, γιατί πολλές φορές ε, το αμελούμε αυτό. Θα πρέπει να δούμε σε τι μέτρα μεταφράστηκαν οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπήρχαν αντισταθμιστικά μέτρα για την άβληση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εφαρμόστηκαν όντω αυτά τα μέτρα. Και οι δημόσιες αρχές, οι δημόσιες αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές έχουν σημαντικό ρόλο εδώ και θα πρέπει να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα. Επίσης, η διαδικασία του κρατικού ελέγχου έχει μεγάλη σημασία για να εξασφαλιστεί διαφάνεια, ποιότητα αλλά και ανεξαρτησία στην κατάρτιση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πολ Κουνάιτ έχει Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε για ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο πρέπει να ομολογήσουμε ότι ε, η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, έχει ακόμα ε, περιπλοκές και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο. Ε, επίσης πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται μεγάλη τεχνογνωσία και πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτοί που αναλαμβάνουν τα σχέδια υποτίθεται ότι έχουν αυτή την πραγματογνωμοσύνη και γι' αυτό ακριβώς τους αναθέτουμε και τα διάφορα ε, σχέδια. Αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει να δικαιολογούνται όλα αυτά τα σχέδια μερικές φορές ε, μπορούν να παρακαμφθούν οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή μερικές άλλες φορές πίσω από τις ΕΠΕ ε, βλέπουμε άλλα πράγματα. Ε, ας πούμε χθες μιλούσαμε για την αρχή της ανεξαρτησίας τα έθνη. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και αυτό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. έχει ο κύριος Λίχτεφριντ για για μισό λεπτό σας παρακαλώ θα παρέμβετε. Κύριε Λίχτεφιρ, μισό λεπτό. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορεί να μην κατάλαβα σωστά τι είπε η συνάδελφο, αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αν υπάρχουν κανόνε, οι κανόνε αυτέ να τηρούνται και να μην ε, είναι παντά σκοπό μα ε, να λέμε «Ε, εντάξει, είναι οι συνθήκε διαφορετικέ, να τα τηρήσουμε επακριβώ. Όχι, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Μήπω εννοούσατε ότι οι κανόνε θα πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από τι συνθήκε και δεν θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στι εκάστοτε συνθήκε. Ε, η κυρία Μολκουνάιτε θέλει να απαντήσει, έχει το δικαίωμα για μισό λεπτό. Θέλετε να απαντήσετε, κυρία συνάδελφε. Σα ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι βεβαίω είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθούμε τους κανόνε όμως. Μερικές φορέ υπάρχουν περιπτώσει ότι κάποιοι, όπου κάποιες ε, ομάδες συμφερόντων προσπαθούν να ασκήσουν πίεση έτσι ώστε ε, να σταματήσουν κάποιο σχέδιο. Ε, αλλά η ανάλυση και η ανεξαρτησία των πραγματογνώμων, πραγματογνωμόνων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό. Και η κυρία Κάντερμπαχ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κάτσου διά έχει ζητήσει. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση καταδεικνύει ότι στο θέμα του περιβάλλοντος έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα πρόβλημα επικοινωνίας συγκεκριμένα. Γιατί ανά πάσα στιγμή μιλάμε για περιβάλλον, για οικονομία, αλλά και είναι αντίθετε αξίε. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα. Χρειαζόμαστε και υποστήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα τη οικονομία. Γιατί νομίζω ότι αυτό δεν το τονίζουμε παρκώ. Τα μέτρα τα οποία ε, προστατεύουν το περιβάλλον, τη φύση, μπορούν να δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας. Γιατί πάντα υπάρχει πόλος τη σήμερα. Είτε φύση είτε θέσεις εργασίας. Και δυστυχώς αυτό και η πολιτική και εμείς ε, χρησιμοποιούμε τα επιχειρήματα αυτά. Θα ήθελα να σας καλέσω να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια συνείδηση προ αυτή την κατεύθυνση, ότι χρειαζόμαστε ανέπαφο περιβάλλον για να υπάρχει οικονομία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ράντσορφ έχει το λόγο. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η, Αυστρία α, καταψήφισε το πυρηνικό εργοστάσιο στον Είναι περίεργη η κατάσταση στην Ευρώπη και νομίζω ότι το πείραμα, το πείραμα αυτό ήταν πολύ δαπανηρό. Για ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με την απάντηση που έλαβα, αλλά ήθελα ένα μόνο στοιχείο να διευκρινίσω. Οι σημερινές προδιαγραφές προβλέπουν ότι οι πίστες σκι μπορούν να υπολογιστούν στις ιοριακές τιμές όταν κατά την δημιουργία της ε, εγκατάστασης προβλέπονται ε, κατασκευαστικές ε, αλλαγές. Όλες αυτές οι εκτάσεις σε διαφορετική περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Θεωρώ ότι η αξιοποίηση μιας επιφάνειας, μιας έκτασης συνεπάγεται την ανάγκη συμπερίληψης της σε τέτοια έργα. Και κάτι άλλο, σε ένα μικρό μέρος ε, κράτους μέλους υπάρχουν δυνατότητες ε, να διακοπεί μια τέτοια διαδικασία. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια δυνατότητα παγώματος. Ε, μπλε κάρτα θέλει να α, α, παρέμβει στο κύριο Βίλαντ. Μισό λεπτό παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Μία ερώτηση προς τον συνάδελφο Βίλαντ που είναι νομικός. Αν και οι ορειβάτες οι οποίοι διασχίζουν τα βουνά που χρησιμοποιούν για παράδειγμα ανελκυστήρες, να τους συμπεριλάβουμε και αυτούς και άλλα άτομα που χρησιμοποιούν ε, διάφορες ε, συσκευές. Χρειάζεται και εκεί μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου να δούμε τα κριτήρια που εννοεί. Ε, ο κύριος Βίλαντ μισό λεπτό για να απαντήσει και τελειώνουμε εδώ τις παρεμβάσεις. Um um για να διευκρινίσω το εξής. Η φύση δεν είναι ιδιοκτησία των ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τον κόσμο. Δεν θεωρώ ότι η συγκεκριμένη περιοχή θα έπρεπε να αποτελεί περίπτωση παγώματος. Κύριε Βίλαντ και σύντομος ήσασταν. Τώρα τη συζήτηση θα κλείσει ο Επίτροπος, ο κύριος Σέτιγκερ. You have the floor, Mr. Commissioner. Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ. Καταρχά, πιστεύω ότι όλοι διαπιστώνουμε ότι η προκειμένη περίπτωση δεν ε, διεξήχθη με τον τρόπο που έπρεπε, με τον δέντε τρόπο αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση εξυπηρετεί το ευρωπαϊκό μας έργο. Διαπιστώσαμε ότι στην συγκεκριμένη υπόθεση οι οριακές τιμές ε, εφαρμόστηκαν με λανθασμένο τρόπο, δεν έγινε το σχετικό screening, ο σχετικός έλεγχος και έτσι δεν ήταν αντικειμενική η εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά δεύτερον, ότι η οδηγία ΕΠΕ στην Αυστρία ε, έπρεπε να προσαρμοστεί να αναθεωρηθεί, προκειμένου να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, με τις δικές σας προδιαγραφές. Κατά τρίτον, είναι σημαντικό τα περαιτέρω μέτρα για τις περιοχές για περαιτέρω έργα να υπάγονται σε ειδικό έλεγχο σε ό,τι αφορά το σύνολο του έργου με τα μεμονωμένα τμήματα του έργου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξετάζουμε ιδιαίτερα και έχουμε ιδιαίτερα στην προσοχή μας την όλη περιοχή. μετά ως Επιτροπή είναι ανοιχτό το κατά πόσο θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία επί παραβάση. Δεν απειλούμε με κάτι τέτοιο, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η δυνατότητα. Εν γέννη, έχουμε και το θέμα της αναθεώρησης της οδηγίας ΕΠΕ. Τι προτείνει ο συνάδελφος Ποτότσνικ. Καταρχάς, να θέσουμε νέους πολιτικούς στόχους. Ε, ποικιλία, βιολογική, ενέργεια, διευρωπαϊκά δίκτυα ε, πολιτική συνοχής. Κατά δεύτερον, να λάβουμε υπόψη τις ε, αποφάσεις του ΔΕΚ, οι οποίες ε, μας οδηγήσαν σε σημαντικές διευκρινήσεις. Τρίτον, το θέμα της βουλευτού Λίχτενμπέργκερ. Διαπιστώσαμε ότι η Αυστρία στο θέμα των οριακών τιμών Παρουσίασε θέματα, σε θέματα ε, διαφάνειας, συμμετοχής των πολιτών, αν υπάρχει επαρκής ε, μεταχείριση από πλευρά των αυστριακών αρχών, αυτό θα το ερευνήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Σε ό,τι αφορά θέματα διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών, θα πρέπει να υποβάλουμε εγγράφως την απάντησή μας και θεωρώ ότι του χρόνου θα καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική επεξεργασία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας βάσει και των όσων μάθαμε από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μας ρωτάτε πώς ε, ορίζεται η επιφάνεια, η έκταση. Θα σας υποβάλουμε γραπτή απάντηση γιατί νομίζω ότι αν εδώ ένας ε, οικοδομηθεί, μάλλον κατασκευαστή ένας ανελκυστήρας, δεν μετράμε μόνο τα τετραγωνικά μέτρα κάτω από τον αναβατήρα. Ούτε μετράμε όμως το σύνορο του βουνού. Υπό τη στενή έννοια, σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η έκταση της πίστας. Και αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συνυπολογιστούν απαραίτητα για τον καθορισμό της οριακής τιμής. Και αυτά θα διευκρινιστούν με σαφήνεια στην οδηγία. Ελέγχοντας τώρα το θέμα το πώς θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε πιο έγκαιρα. Γιατί όντως εδώ πλέον ερχόμαστε πέντε χρόνια μετά την απόφαση ε, κατασκευής. Ερχόμαστε καθυστερημένα. Υπάρχει όμως επικορικότητα και η ευθύνη για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών ε, προτύπων καταρχάς εναπόκειται στα χέρια των κρατών μελών. Θεωρώ ότι ιδιαίτερα στην Αυστρία λόγω της ε, υπόθεσης αυτής θα υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα τέτοια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, η συζήτηση, τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, έληξε εδώ. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα παραπλανητικές πρακτικές των εταιριών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων. Ξεκινάμε με τις